ημερήσια διάταξη έχει δημοσιευτεί στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ τους υπαλλήλους και τους διερμηνείς που μας συνόδευσαν μέχρι αυτή την